της κοινοβουλευτικής του ασυλίας και αυτό το αίτημα θα παραμευθεί στην Αρμόδια Επιτροπή. Από τις ομάδες του Κοινοβουλίου και τους μη εγγεγραμμένους έχουμε αιτήματα για ορισμούς στις διάφορες επιτροπές και αντιπροσωπείες. Αυτά έχουν δημοσιευτεί. Εάν μέχρι τη δημοσίευση των πρακτικών δεν έχουν υπάρξει αντιρρήσεις, θεωρούνται πως εγκρίνονται. Η κυρία Αγγέλικα Βέρτμαν μου ανακοίνωσε πως προσχώρησε στην ομάδα των φιλελευθέρων. Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου